Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά το Κοινοβούλιο λειτουργεί βάσει διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων και νομίζω ότι όλα τα πολιτικά δόγματα έχουν το ίδιο δικαίωμα να συμμετέχουν για την εξέβρεση μιας κοινή λύσης. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει το προνόμιο να πει ότι κάποια πολιτική πεποίθηση δεν είναι ε, σωστή και δεν αξίζει να συμμετέχει στην κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, κύριοι βουλευτές και κυρίες βουλευτές για την ε, ακρόαση αυτή, τον κύριο Μοσκοβίση για τις απαντήσεις σου και τώρα θα σας καλέσω να κάνετε ένα καταλεκτικό, μια καταλεκτικά σχόλια μέχρι πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχήν ευχαριστώ για την ανταλλαγή αυτή. Ήταν ειλικρινείς, άμεσες και απαιτητικές οι ερωτήσεις και στο σεβασμό, με σεβασμό στις γλώσσες μας και στις παραδόσεις μας και να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία τους διερμηνείς που μας βοηθούν στην άσκηση της πολυγλωσσίας. Ελπίζω ότι σας απήντησα όσο γινόταν καλύτερα να καταλάβατε την ειλικρίνειά μου, τις ευρωπαϊστικές μου επεπιθήσεις και ε, ότι θα μπορέσω να καταφέρω εις πέρα στα καθήκοντα που, για τα οποία είμαι υποψήφιος. Θα ήθελα τέλος να σας αναφέρω ποιες είναι οι επιθύσεις μας, οι επιθύσεις που θα καθοδηγήσουν την εργασία μου τα επόμενα πέντε χρόνια, αν βεβαίω με επικυρώσετε. Καταρχήν θα έχω την ευθύνη αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Με αυτό το γενικό ε, κοινό ε, συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ιδεώδε, είναι ένα, προ, ένα πρότυπο. Ε, από, οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, όπω έλεγε ο Ζακ Τελόρ, και ένα σύνολο κανόνων επίση. Να ζήσει το ευρωπαϊκό πνεύμα, θα, θα μεριμνήσω και να ευημερήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο. Και οι κοινοί κανόνε θα είναι η πηξίδα μου, η μόνη μου πηξίδα. Ω Ευρωπαίο Επίτροπο θα ε, ε, ενεργήσω με βάση τι επιλογέ του Προέδρου Jean-Claude Juncker. Αυτό σημαίνει ότι μαζί θα χαράξουμε σαφεί προτεραιότητε, να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη τη υπήρου μα, ε, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, να καταπολεμήσουμε τι ανισότητε, να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, τη φοροαπάτη, να ενεργήσουμε κατά τον τραστ, διαφάνεια, να προστατεύσουμε κυρίω χάρη στα Δελανία του συμπολίτε μα από τι υπερβολέ τη παγκοσμιοποίηση αυτέ. Οι προτεραιότητε που είναι προτεραιότητε του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ είναι και θα είναι και δικέ μου. Ω Ευρωπαίο Επίτροπο ε, θα οδηγούμε από το πνεύμα τη ομαδικότητα και η νέα οργάνωση που προτείνει ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ με βρίσκει απολύτω σύμφωνο. Δεν πρόκειται για εποπτεία, ιεραρχία και δαιμονία. Οργανώνεται μια ειδική ε, και πρωτότυπη ε, απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων από πλευρά του Προέδρου. Ε, οφείλουμε όλοι έτσι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε και μέσα στην ομαδικότητα, στο ομαδικό πνεύμα θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους επιτρόπους και αντιπροέδρους και κυρίως με τους δύο αντιπροέδρους με τους οποίους θα είμαι σε ομάδα καθημερινά τον κύριο Ντομπρόφσκι και τον κύριο Κατάινεν. Να σας το πω ξεκάθαρα, μεταξύ των τριών μας δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός τεχνητής φύσης. Δεν μπορεί να υπάρχει γραφειοκρατικός ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικές διαφορές οι οποίες να ε, κυριαρχούν επί των υπολείπων θεμάτων. Γιατί αν δεν το καταφέρουμε αυτό θα χάσουμε ενέργεια, χρόνο που θα ζημιώσει τα όσα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Οφείλουμε και θα είμαστε μια ομάδα ενωμένη γύρω από τους ίδιους στόχους. Και σε αυτό δεσμεύομαι, το έχω συζητήσει μαζί τους, ξέρω πως είναι και το δικό τους πνεύμα το ίδιο. Και τέλος, ως Ευρωπαίος Επίτροπος, θα συνεργαστώ στενά με το Ευρωκοινοβούλιο και καταρχήν με το μέλη των επιτροπών σας. Και για μένα αυτό δεν είναι λόγια του αέρα επειδή τώρα βρίσκομαι εδώ. Είναι βαθύτατη μου πεποίθηση. Πριν από ακριβώς 20 χρόνια μπήκα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είδα να μεγαλώνει, να αλλάζει, να γίνεται πραγματικός συνομοθέτης και εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών λαών. Εσείς είστε εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Εσείς ενσωματώνετε την δημοκρατική νομιμότητα, εκλέγεστε με καθολική ψηφοφορία και αυτό μας αναθέτει κοινέ ευθύνε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων πέντε ετών στην Ευρώπη. Και αυτό ήθελα να σας πω. Απάντησα στις ερωτήσεις σας, κάποιες φορές ήταν δύσκολες. Το έκανα χωρίς ε, ε, φτιασίδια, ε, ειλικρινά. Είμαι έτοιμος να συνομιλήσω μαζί σας, να είμαι σε διάλογο μαζί σας για να έχουμε αποτελέσματα στην Ευρώπη. Επ' αυτόν θα κριθούμε. Και εσείς και εγώ και όλη η Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτές, κύριε Πρόεδρε, το να γίνω, υποψήφι, να γίνω επίτροπος με συγκινεί, γιατί είναι για μένα τιμή και είναι και μια, ένα ένδοξο ε, βήμα στην πορεία μου, στις ευθύνες που έχω αναλάβει, αλλά βεβαίως με σοβαρότητα προσεγγίζω αυτή την καταξίωση ε, είμαι, έχω τις πεπιθήσεις μου και ε, ελπίζω να σας έπεισα για την ισχύ της εμπειρίας μου, την ισχύ της δέσμευσής μου, της ανεξαρτησίας μου και της βούλησής μου να συνεργαστώ θετικά μαζί σας. Σας ευχαριστώ για τις τρεις ώρες αυτές που περάσαμε μαζί. I would like to thank you. Πρόεδρος, να σας ευχαριστήσω κύριε υποψήφιε επίτροπε για τη σημερινή σας εμφάνιση εδώ σε αυτή την ακρόαση και για την επιθυμία σας να μπείτε στην πλούσια αυτή εντατική και καρποφόρα νομίζω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες θα γίνει συνεδρία των επιτροπών και κλεισμένων των, θυρών, των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών από τη μία μέχρι τις δυόμιση. Σας ευχαριστώ. Τέλος συνεδρίασης.